παρατηρήσεις επί της ουσίας, έτσι ώστε από κοινού να καταστούμε όλοι πλέον αποτελεσματικοί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπερές. Έτσι θα κλείσουμε τη συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12 το μεσημέρι. Πάμε στο επόμενο σημείο της σημερινής τη διάταξης που είναι η κοινή συζήτηση σε σχέση με τα χρηματοοικονομικά εργαλεία. Δεν θα σας αναγνώσω τον κατάλογο των εργαλείων. Και προσκαλώ τον πρόεδρο της αντιπροσωπείας συνδιαλλαγής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Βιδάλ Κουάδρας, να λάβει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Στο πολύ κύριε Πρόεδρε. Μετά από μακρές και εργώδεις διαπραγματεύσεις, η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτή τη διαδικασία συνδιαλλαγής ενέκρινε τη συμφωνία η οποία επετεύχθη με το Συμβούλιο με ευρεία πλειοψηφία στις 25 Οκτωβρίου. Στην αρχή της παρεμβασή μου θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς όλους τους συναδέλφους από την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ιδίω αυτού που βρίσκονται στην ομάδα διαπραγμάτευση και στο Συμβούλιο για την ανοιχτή του στάση και προ την Κομισιόν τη μόνιμη βοήθεια που μα έδωσε. Πρέπει να πω, ως πρόεδρος αυτής της Επιτροπής Διαλλαγή ότι το αποτέλεσμα στο σύνολό του πρέπει να θεωρηθεί ικανοποιητικό για το Ευρωπαϊκό Κοινόβουλιο. Είχαμε μπροστά μα μια πολιτική πρόκληση, μια πρόκληση η οποία ήταν και από πνευματική άποψη σημαντική και ενδιαφέρουσα να προσαρμόσουμε τα δημοσιονομικά μας εργαλεία στις απαιτήσεις της νέας συνθήκης. Και αυτό επετέχθη κύριε Πρόεδρε με το να εγγράψουμε τις ουσιαστικές πτυχές αυτών των εργαλείων, τις προτεραιότητες, τους στόχους, τα αποτελέσματα τα οποία προσδοκούμε και την κατανομή των πόρων σε πραγματικούς όρους, να τα εγγράψουμε όλα αυτά στο πλαίσιο της συναπόφασης. Έτσι θέτουμε το Συμβούλιο αλλά και το Κοινοβούλιο σε επίπεδο απόλυτης ισορροπίας, ισότητος. Χάρη σε αυτές τις συζητήσεις μπορώ να σας πω ότι η Κομισιόν μπόρεσε να ενισχύσει ιδιαίτερα την δήλωσή της σε σχέση με την χρήση των κατεξουσιοδότηση πράξεων στα μελλοντικά χρηματοοικονομικά εργαλεία Και ένα άλλο σημείο το οποίο θέλω να υπογραμμίσω είναι η πολιτική δήλωση του Συμβουλίου σε σχέση με τη χρήση των κατεχώρησης κατεξουσιοδότηση πράξεων σε ε, περιπτώσεις όπου το Συμβούλιο είναι δεσμευμένο να θεωρήσει ότι θα είναι <clears throat> έγκυρες αυτές οι θέσεις. Εκεί ήταν μια κόκκινη γραμμή του Συμβουλίου όπου αντιστάθηκε. Τελικά το εδέχθη όμως. Για τα ίδια τα εργαλεία αυτά. Στην περίπτωση του εργαλείου για τις ε, βιομηχανικές χώρες καταφέραμε σε ένα παράτημα να αναφέρονται τα κατόφλια των πόρων κατά γεωγραφική περιοχή και κατά τομής. Στο ε, μέσο για τις χώρες που εξάγουν μπανάνες. Επίσης καθορίσαμε τον τρόπο κατανομής των πόρων και τη μεθοδολογία η οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί και έτσι εξαλείψαμε οποιαδήποτε αυθαίρετη φύση ή οποιοδήποτε περιθώριο ελιγμών για την Κομισιόν που να μην υπόκειται στον έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρέπει να πω ότι <clears throat> ένα συγκεκριμένο στοιχείο σε αυτό το μέσο δεν κατάφερε το Κοινοβούλιο να ε, σε αυτό το σημείο να περάσει τη δική του θέση. Αλλά κύριε Πρόεδρε, μία συνδιαλλαγή είναι συμφιλίωση θέσεων. Δεν μπορεί να την κερδίσει κανείς κατά 100%. Όπως λοιπόν θέσαμε και εμείς τις κόκκινες γραμμές μας και το Συμβούλιο μπορούσε να έχει κόκκινες γραμμές. Θέλω να προσθέσω κύριε Πρόεδρε ότι εάν δεν εγκριθεί από το Κοινοβούλιο αύριο το μέσο αυτό το οποίο αφορά τις χώρες οι οποίες είναι εξαγωγής μπανάνας, το αποτέλεσμα θα είναι πολύ σοβαρό. Αυτή η απόφαση θα έχει πολύ σοβαρό χαρακτήρα και πολλές συνέπειες. Τα προγράμματα αυτά θα ακυρωθούν και αντίθετα από ό,τι λένε ορισμένοι συνάδελφοι που πιστεύω το λένε καλή την πίστη. Δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχουν κονδύλια σε άλλες περιοχές του προπολογισμού για να υποστηριχθούν αυτά τα προγράμματα. Επομένω, <clears throat> ιδιαίτερα ευάλωτοι κοινωνικοί τομή σε αυτές τις χώρες θα πληγούν από την απόφασή μα και οι πολιτικές συνέπειες θα είναι πάρα πολύ βλαβερές. Και θα έχουν και επίπτωση στις συμφωνίες μας στον ΠΟΕ, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, για τις μπανάνες που και αυτές θα διαταραχούν. Θα διαταραχθούν. Κλείνω λέγον κύριε Πρόεδρε. Το Συμβούλιο ενέκρινε ήδη αυτή τη συμφωνία, ώστε με τη συμφωνία κυρίων που έχουμε επιτύχει με το Συμβούλιο, ελπίζουμε ότι αύριο θα μπορέσουμε να είμαστε συνεκτικοί και θα εγκρίνουμε αυτή τη συμφωνία. Έτσι, η δική μου σύσταση ως Πρόεδρου της Επιτροπής Συνδιαλλαγής, κύριε Πρόεδρε, είναι αύριο να δώσει την υποστήριξη του Κοινοβούλιο σε αυτή τη συμφωνία συμφιλίως. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστώ πολύ και τώρα οι εισηγητές. Ο κύριος Γκέρενς πρώτος. Τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Οι κανονισμοί που αφορούν τα συνοδευτικά μέτρα στο τομέα τη παράνοση έχουν δύο πτυχέ. Ο, ο ένας, η μία πτυχή έχει θεσμικό χαρακτήρα και, και άλλη αφορά την χρηματοδότηση. Ο θεσμικό χαρακτήρα αφορά τη συναπόφαση στο Κοινοβούλιο. Για την, για την άλλη πτυχή δεν υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή ω προ τι θεσμικέ πτυχέ υπάρχουν τα προβλήματα και εδώ έχουμε σημαντικέ αποκλήσει. Πώ μπορούμε δηλαδή να καταστήσουμε τον κανονισμό Μπάμα, συνοδευτικά μέτρα Μπανάνα δηλαδή, ε, σύμφωνο με το με τη συνθήκη της Λισαβόνας και δει το άρθρο 290 αυτής συγκεκριμένα τη συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπεται πως το Κοινοβούλιο έχει ισότιμες με το, κοινό, με το Συμβούλιο Εξουσίας όσον αφορά την έγκριση των στρατηγικών προτεραιοτήτων για τον προγραμματισμό των ευρωπαϊκών μέσων συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν στην αναπτυξιακή συνεργασία. Ως εισηγητής και με βάση και την εντολή που έχει προσδορίσει η διάσκεψη των Πρόεδρων του Κοινοβουλίου και δυνάμει και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί και σε επίπεδο Επιτροπή Ανάπτυξη ε, και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την αντιπροσωπεία του στην ε, συνδιαλλαγή. Στου οκτώ τριμερεί διαλόγου με το Συμβούλιο και την Επιτροπή ακολούθησα τι δύο εξή κόκκινε γραμμέ. Πρώτον, δεν υπάρχει περίπτωση να παραιτηθούμε από την ισότιμη μεταχείριση Συμβουλίου Κοινοβουλίου προ τον προσδορισμό των προτεραιοτήτων για τον χρηματοπιστικό προγραμματισμό δημοσιονομικό προγραμματισμό και στο δεύτερο δεύτερη κόκκινη γραμμή δεν υπάρχει περίπτωση να υποχωρήσουμε ως προς τον ε, δημοκρατικό έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην υπόθεση αυτή, πράγμα το οποίο θα αποτελούσε ένα πολύ αρνητικό προηγούμενο. Μετά τους, αυτούς, τους 8 αυτούς τριμερείς διαλόγους και την πολύ δυσάρεστη στάση που ακολούθησε το Συμβούλιο, το οποίο δεν είναι καν παρόν εδώ, έχουμε δύο διαφορετικές αντιδράσεις. Αφενός μεν η αντιπροσωπεία στην πλειοψηφία της υπερψηφίζει τη συμβαστική πρόταση που σας έχει υποβληθεί, πλην όμως μια ισχυρή μειοψηφία δεν εγκρίνει την προτινόμενη συμβαστική πρόταση στο πλαίσιο τη διαλλαγή. και έτσι ως ε, εκπρόσωπος ε, της αντιπροσωπεία, ω εισηγητής δηλαδή, αλλά και σεβόμενος στη Δημοκρατία, είμαι υποχρεωμένος να σας ε, αποδώσω τα αποτελέσματα αυτών των εργασιών. Η δική μου ερμηνεία της κοινοβουλευτική διοντολογία θα μου απαγόρευε να αποκρύψω τα δεδομένα αυτά, τη διαφοροποίηση αυτή δηλαδή. Ταυτόχρονα όμω, η ίδια αυτή η δημοκρατική διοντολογία μου, ε, με, με υποχρεώνει να δηλώσω ότι δεν είναι ικανοποιητικά τα αποτελέσματα καθόλου. Και γιατί δεν είναι, διότι σε περίπτωση έγκρισης αυτής της πρόταση από το Κοινοβούλιο μπορεί να αποτελέσει αυτή πολύ δυσάρεστο προηγούμενο, πολύ κακό προηγούμενο στο πλαίσιο δηλαδή του σχεδίου BAM, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει μόνο δικαίωμα για ενημέρωση ω προ τι στρατηγικέ επιλογέ τι οποίε θα προφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο θέμα τη ε, ε, καταχώρηση αυτών των πιστώσεων των 190 εκατομμυρίων ευρώ. Μόνο ενημέρωση λοιπόν το Κοινοβούλιο και έτσι το Συμβούλιο θα, είναι μόνο το αρμόδιο, ε, θα έχει μόνο την εξουσία να αποφασίσει με βάση προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό δεν αποτελεί λοιπόν βήμα προ τα εμπρό. Αλλά δύο βήματα οπισθοδρόμηση. Ένα βήμα οπισθοδρόμηση προ τη συνθήκη τη Λισαβόνα και δεύτερο βήμα οπισθοδρόμηση σε σχέση με την κατάσταση που ίσχυε πριν από την 1η Ιανουαρίου του 2009, κατά την ημερομηνία αυτή που ξέρετε, θα τέθησε ισχύ η συνθήκη τη Λισαβόνα. Μέχρι το 2009 δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο μια λεγόμενη αρνητική διαδικασία και τη δυνατότητα να έρθει σε αντιπαράθεση με τι θέσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με ανασταλτικό χαρακτήρα η διαδικασία. Τώρα όμω πλέον δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα και το Συμβούλιο έχει καταφέρει να αποστερήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι συνομοθέτη όμω, μαζί με το Συμβούλιο, το δικαίω, του δικαιώματό του για το δημοκρατικό έλεγχο. Αποδεχόμενο μόνο αυτό το Συμβούλιο ε, να μπορεί, τη λύση μόνο αυτό το Συμβούλιο να μπορεί να εγκρίνει τα μέτρα εφαρμογής ε, του κανονισμού ΜΠΑΜ. Δηλαδή με μια πολύ ειδική ερμηνεία του άρθρου 291 και έτσι βλέπουμε δύο βήματα οπισθοδρόμησης. Γι' αυτό δεν μπορώ να υπερψηφίσω την έκθεση. Αλλά αποδέχομαι ότι πρόκειται για μια πολύ δύσκολη προσωπικά απόφαση, την οποία όμως λαμβάνω με τα λόγω γνώσης γιατί θεωρώ ότι δεν μπορούμε να προδικάσουμε έτσι και να προκαταλάβουμε περαιτέρω διαδικασίες διαπραγμάτευσης και συνδιαλλαγή για τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Σας ευχαριστώ πολύ και το δίνω το λόγο στον κύριο Σόλτσε για τέσσερα λεπτά. Ε, πρόεδρε, Επίτροπε, συνάδελφοι, όταν έλαβα το φάκελο αυτό δεν είχα υπολογίσει ότι θα με απασχολούσε εντατικότατα μάλιστα επί δύο χρόνια και πλέον. Θεωρώ ότι στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι δύσκολο να το μεταβιβάσουμε αυτό και να το εξηγήσουμε. Ιδιαίτερα επειδή μπορούσε να επιτευχθεί ε, συνεννόηση μέσα σε λίγους μήνες σε ό,τι αφορά την ερμηνεία της ε, συνθήκης της Λισαβόνας και της ερμηνείας των κατά πράξεων αποτελεί την αιτία και η άρνηση των κρατών μελών, σε κάποιων κρατών μελών, να δώσουν περισσότερες αρμοδιότητες ελέγχου στο Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο είχαν συμφωνήσει ότι το χρηματοκεντρικό μέσο θα έπρεπε να αλλάξει για τις εκβιομηχανισμένες χώρες και θέλαμε να απελευθερώσουμε ένα μεγάλο ποσό μέχρι 176 εκατομμύρια ευρώ για το Erasmus ε, Mundus, για πολιτισμό, προτιμ... ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το καθεξής. Ε, οι μικρές, μικρομεσαίες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα ωφελούνταν από τη διαδικασία αυτή. Αλλά η καθυστέρηση είχε ως αποτέλεσμα να είναι πολύ πιο περιορισμένο το ποσό αυτό επενδύσεων στις τρέχουσες δημοσιονομικές προοπτικές. Γι' αυτό μας λυπεί ιδιαίτερα γιατί θα μπορούσαν, μπορούν να επενδύονται ε, χρήματα και δαπάνε σε αναπτυσσόμενες χώρες και μάλιστα θα ήταν project αυτά τα οποία θα, δεν θα επίπταν στον κανονισμό για τις αναπτυσσόμενες χώρες όπως για παράδειγμα σε χώρες όπως η Ασία και η Λατινική και οι περιοχές όπως η Λατινική Αμερική μέσω της γεωγραφικής αυτής ε, επεκτάσεων θα μπορέσουμε να δώσουμε πιο πολλές ευκαιρίες. Ε, θα έπρεπε να είναι σαφές όμως για ποιον σκοπό θα, θα χρησιμοποιούνται τα επιπλέον αυτά κονδύλια. Στο παράρτημα 2 απαριθμούνται αναπτυσσόμενες χώρες και 5% των ε, πόρων δαπανούνται για διπλωματία. για αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω η δημοκρατία και ο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 20% για την προώθηση άμεσων σχέσεων μεταξύ των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των χωρών εταίρων. Επίση, έμφαση στην ακαδημαϊκή ε, εκπαίδευση και στην ε, δικτύωση των ε, φοιτητών και 50% των πόρων δαπανώνται για την δικτύωση επιστημονικών κοινοτήτων, όπου επίκεντρο, στο επίκεντρο βρίσκονται πάλι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και εστιαζόμαστε σε χώρες ε, οι οποίες στηρούν τις, ε, τα πρότυπα της Παγκόσμιας Οργάνωσης ε, Εργασίας και που συγκεντρώνονται στην μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Και για τα πρακτικά και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το μέσο αυτό δεν πρέπει να αποτελέσει κρυφή επιδότηση τηλεφωνικών υπηρεσιών και εταιριών στην Κολομβία ή σε, άλλον σε άλλες ε, χώρες της Λατινικής Αμερικής. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να φροντίσουμε να τηρηθούν οι βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς συμβιβασμούς, γιατί στο μέλλον θα πρέπει να υπάρχει και συνοχή στις πολιτικές των ε, αναπτυσσόμενων χωρών. Εμείς ως Κοινοβούλιο δεν θα πάψουμε να ελέγχουμε τα στοιχεία αυτό. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει ειδική ε, υποχρέωση αναφοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τον κανονισμό αυτό. Θέλουμε να ελέγξουμε κατά πόσον η πολιτική ε, σχεδιασμός ανταποκρίνεται στο πνεύμα των άλλων χωρών. Γι' αυτό λοιπόν θα, θέλουμε να, θα θέλαμε να ε, καθιερωθούν και να αναγνωριστεί η σημασία των ε, πράξεων κατά εξουσιοδότηση και το δικαίωμα του ΒΕΤΟ. Με το μέσο αυτό, όπως και με όλα τα άλλα μέσα, και συμφωνώ και με τον εισηγητή, θα ενισχύσουμε και θα προασπίσουμε τα δημοκρατικά αυτά δικαιώματα για το μέλλον. Ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Γκάλα έχει το λόγο. Τα Ευχαριστώ, Πρόεδρε. αξιότιμη Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Οι συνάδελφοί μου ήδη ανέφεραν ότι όλοι μείναμε έκπληκτοι που οι διαπραγματεύσεις προκάλεσαν τόσο μεγάλες αντιδράσεις και τόσο μεγάλη αντίσταση κατά το δικαιώματο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ασκεί δημοκρατικό έλεγχο. Όλοι μείναμε έκπληκτοι που τράβηξαν τόσο σε μάκρο οι διαπραγματεύσει, γιατί κανένα από του συζητητέ δεν είχε φανταστεί ότι θα έπαιρνε τόσο χρόνο οι διαπραγματεύσει. Παρ' όλα αυτά, χαίρομαι που σήμερα εδώ ε, κάνουμε την τελική συζήτηση για τα θέματα αυτά, προκειμένου και να ολοκληρωθούν στην έκθεση για το χρηματοδοτικό μέσο για την πραγωγή της δημοκρατίας εργάστηκα και θα ήθελα να τονίσω ότι το μέσο αυτό σκοπό έχει να προάγει την δημοκρατία και τα ε, δικαιώματα, των ανθρώπινα δικαιώματα. Μιλάμε για την καταπολέμηση της αντικής ποινή και όλα αυτά υποστηρίζουν και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις που δραστηριοποιούνται προς αυτή την κατεύθυνση στις τρίτες χώρες. Τα διδάγματα της Αραβικής Άνοιξης μας έχουν δείξει πόσο σημαντικό είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετέχει στη διαμόρφωση των στρατηγικών αυτών ζητημάτων και ασφαλώς είναι πάρα πολύ σημαντικό σημαντική, πολύ σημαντικό πώς δαπανούνται τα κονδύλια του χρηματοδοτικού μέσου. Από την πρώτη ανάγνωση πετύχαμε ε, συμφωνία σε ό,τι, αφορά, σε αφορούσε το περιεχόμενο. Θέλαμε να υποστηριχτούν οι μη κυβερνητικέ οργανώσει σε επιτόπου. Στις ε, δύο επόμενε αναγνώσει, το θέμα ήταν το ελεγκτικό δικαίωμα, τα δικαιώματα ελέγχου, οι αρμοδιότητε ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ήταν μια συμβολική στιγμή, θα έλεγα, γιατί στο σημείο αυτό έπρεπε να φανεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την 1η Δεκεμβρίου του 2009 έλαβε νέο και πιο μεγάλο ρόλο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Βιντεγάλ Κουάντρας και όλους όσοι συμμετείχαν στον αγώνα αυτό τους τελευταίους μήνες. Όλοι γνωρίζουμε ότι ήταν μακρύς ο δρόμος και γνωρίζουμε επίσης ότι σε ένα συμβιβασμό πάντα και τα δύο μέρη πρέπει να προσεγγίσουν το ένα το άλλο. Παρ' όλα αυτά, έχω την αίσθηση ότι καταφέραμε να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα προς το εμπρός. Και είναι ιδιαίτερη επιτυχία το γεγονός ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο στο μέλλον θα καθορίζουν την, τον στρατηγικό σχεδιασμό από κοινού. Και είμαι πεπισμένη ότι η συμφωνία η οποία προέκυψε θα ενισχύσει την διαπραγματευτική θέση του Κοινοβουλίου στο μέλλον είναι πραγματικά εξαιρετικά σημαντικό σε θέματα δημοκρατίας, σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις ε, χώρες αυτές. Το θέμα όμως δεν είναι μόνο η εμπιστοσύνη μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά ε, τέτοια θέματα, αλλά το θέμα είναι και η ευθύνη μας έναντι των χωρών του τρίτου κόσμου. Γι' αυτό λοιπόν σα παρακαλώ να υπερψηφίσετε αύριο αυτά τα τέσσερα χρηματοδοτικά μέσα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ. Και τώρα παρακαλώ την κυρία Λόχμπιλερ να λάβει το λόγο. Τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Όσο συνεισυχητρία αυτής της έκθεσης θα ήθελα και εγώ να πω δύο λόγια για το περιεχόμενο. Οι αλλαγέ που παρουσίασαν στο φυστάμενο μέσο δίνουν τη δυνατότητα κατά εξαίρεση να καλυφθούν δαπάνες που σχετίνονται με τέλη που καταβάλουν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις όταν συμμετέχουν σε προγράμματα και σχέδια και έργα, πράγμα το οποίο επιτρέπει καλύτερη ευελιξία στο μέσο, δεδομένου ότι ορισμένε κυβερνήσει πλέον δεν αποκλείουν τι μη κυβερνητικέ οργανώσει από την καταβολή τελών ή φόρων. Και μερικέ φορέ μάλιστα με τον τρόπο αυτό ε, επιβάλλουν περισσότερη πίεση και περιορίζουν το πεδίο δράση του. Πρέπει να πω βεβαίω ότι είναι πάρα πολύ ανησυχητική αυτή η τάση, αλλά και πάρα πολύ πραγματική. Γι' αυτό είναι καλό το ότι μπορέσαμε να επιτύχουμε αυτή την αλλαγή. Επίση, θεωρώ ότι έχει εξασφαλιστεί θετική έκβαση από τη συνδιαλλαγή για το μέλλον τη Δημοκρατία και τη προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την περίοδο 14 με 20 και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε σύντομα μία πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ως αποτέλεσμα αυτών των διαπραγματεύσεών μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει μάλιστα σε μια ανακοίνωση για τον προϋπολογισμό 2020 και παραθέτω ότι η μελλοντική νομική βάση για τα διάφορα μέσα θα προτείνει εκτεταμένη χρήση πράξεων κατά εξουσιοδότηση για να εξασφαλίσει την περισσότερη ευελιξία στη διαχείριση των πολιτικών κατά την χρηματοπιστωτική περίοδο κατά τη δημοσιονομική περίοδο, ε, τηρουμένων βεβαίως ε, και των αρμοδιοτήτων των ε, δύο συναρμόδιων σκελών του προϋπολογισμού. Επίσης, συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο η χρήση των καταξουσιοδότηση πράξεων σε εξωτερικές σχέσεις για το μέλλον στα χρηματοπιστωτικά μέσα, πράγμα το οποίο ενισχύει και την διαπραγματευτική θέση του Κοινοβουλίου στο μελλοντικό μέσον για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε με το Συμβούλιο μας επιτρέπει να επικεντρωθούμε από κοινού στις στρατηγικές, στις προτεραιότητες οι συνδεκτικές ε, κατανομές ποσών και τα αποτελέσματα που θέλουμε. Δηλαδή θα μπορεί το Κοινοβούλιο να έχει περισσότερη παρέμβαση στα κονδύλια που θα θέλει να αποδώσει για τις προτεραιότητες αυτές, για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στα μελλοντικά μέσα. Στο παρελθόν, παραδείγμα, το Κοινοβούλιο διαμαρτύρονταν ότι δεν υπήρχε επαρκή χρηματοδότηση για τις δραστηριότητες ε, σχετικές με τη δημοκρατία και συμπεριλαμβανομένων και των μέσων για τα κοινοβούλια. Τώρα όμως με τις κατεξουσιοδότητε συμπράξει, το μελλοντικό χρηματοπιστωτικό μέσο θα έχουμε περισσότερη ευελιξία για να μπορούμε να αλλάζουμε και προτεραιότητες. Η κατεξουσιοδότηση πράξη θα, θα μας επιτρέπουν να παρεμβαίνουμε όχι μόνο κατά τη γένεση του μέσου, δηλαδή την διατύπωση του κανονισμού όπως τώρα, αλλά και στην, στα έγγραφα πολιετού στρατηγικής. Έτσι, σε τακτικά χρονικά ε, σημεία της διάρκεια αυτού του μέσου θα μπορούμε να παρεμβαίνουμε. Εν τέλει, ναι, δεν καταφέραμε όσα θα θέλαμε σε αυτό το γύρο των διαπραγματεύσεων, αλλά αυτό ενίσχυσε την αποφασιστικότητά μα για το προσεχή γύρο που θα ξεκινήσει από τον Ιανουάριο. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Και τώρα... Στρέφομαι στον τελευταίο εισηγητή ομιλητή, τον κύριο Μίτσελ, για τέσσερα λεπτά. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η διαδικασία συνδιαλλαγής ε, οδήγησε σε κάποια κέρδη, σε κάποια από τα σημεία που ενδιαφέρουν το Κοινοβούλιο Προαλλιότερα υπήρχαν πολλέ ερωτήσει όσον αφορά το βαθμό αρμοδιοτήτων που δίδεται στην Κομισιόν για την εφαρμογή των προγραμμάτων ε, σε σχέση με τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα τη Ένωση. Και είμαι ευτυχή γιατί τώρα η κατάσταση το ε, σημαίνει το Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζουν από κοινού σε σημαντικέ ε, στρατηγικέ αποφάσει και αυτό είναι πολύ θετικό. Οι διαπραγματεύσει ήταν εξαιρετικά δύσκολε και περίπλοκε, ιδιαίτερα αφού το Συμβούλιο δεν ήταν δραστήριο και δεν έκανε ούτε μια αντιπρόταση στις ε, συζητήσεις. Γι' αυτό το Κοινοβούλιο αναγκάστηκε να κινηθεί και να κάνει υποχωρήσεις προς το συμφέρον των χωρών δικαιούχων. Πολλοί από τους ε, ε, συναδέλφους στην Επιτροπή και τους συνεισηγητές θεωρούν ότι αυτός ο κανονισμός ΜΠΑΜ δεν είναι αποδεκτός από, νομικό, από νομική άποψη και θα επιστρέψω στο θέμα αυτό σε λίγο. Εγώ θεωρώ πως ε, τα μέλη του ΕΛΚΑ αποδίδουν μεγάλη σημασία στο δεύτερο τμήμα του σχεδίου νομοθετικού προπολογισμού για τον κανονισμό ΜΠΑΜ. Ε, και ιδιαίτερα στη τελευταία φράση του που λέει και παραθέτω υπογραμμίζει ότι αυτός ο κανονισμός δεν αποτελεί προηγούμενο για τις μελλοντικέ διαπραγματεύσει για την περίοδο μετά το 2013 και τα σχετικά χρηματοδοτικά μέσα. Το Κοινοβούλιο απαιτεί σεβασμό αυτού του όρου σε όλες τις μελλοντικέ διαπραγματεύσει. Ε, αν δεν τηρηθεί αυτή η ρήτρα, το Κοινοβούλιο θα, θα χρησιμοποιήσει τις, ε, τις αρμοδιότητες του επί ελέγχου για πολλές πολυετής στρατηγικές και το βασικό ζήτημα της δημοκρατικής ε, λήψης αποφάσεων και η συνθήκη της αγώνας είναι οι βασικές αρχές για αυτό το θέμα και γι' αυτό και ε, υπογραμμίζω τις ανησυχίες που εξέφρασε και ο κύριος Γκέρος και θα το πω την παρουσία σας κύριε Αντιπρόεδρε είναι πλέον καιρός ο πρόεδρος αυτού του κοινοβουλίου να καλέσει ε, να γίνει μια ανεξάρτητη ε, ε, έρευνα για το ρόλο που πρέπει να παίζει η Κομισιόν ως τίμιος διαμεσολαβητής της διαπραγματεύσεις. Δεν θα πρέπει να παίρνει το μέρος οποιοδήποτε θεσμικού οργάνου. Θα πρέπει να εξασφαλίζει πως οι αρχές που ορίζονται από τις συνθήκες που προς το συμφέρον των ευρωπαϊκών λαών θα τηρούνται όπως άλλωστε είναι και το καθήκον της. Έχω αμφιβολίες για το ότι το πράττει αυτό αυτή τη στιγμή. Τώρα, 36 εκατομμύρια παιδιά πέθαναν παλιότερα. Την ημέρα, ε, χάρη στα προγράμματά μας, αυτός ο αριθμός έχει μειωθεί, έχουμε φτάσει στα 31 εκατομμύρια. Όμως ο πληθυσμός του κόσμου έχει αυξηθεί κατά 2 δις το 90% των οποίων ε, ζουν στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Θα πρέπει λοιπόν να αναπτυχθεί αυτό το μέσο για αλτρουιστικούς λόγου, αλλά και για εγωιστικούς λόγου, γιατί διαφορετικά τα παιδιά μα και τα εγγόνια μα θα έχουν μια φρικτή κληρονομιά. Θα πρέπει να, να καλλιεργήσουμε την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, ε, ξεκινώντα από του ευρωβουλευτέ και του εθνικού βουλευτέ, όσον αφορά τη σημασία τη συνέχιση αυτή τη ε, πορεία. Χρειάζεται συνοχή, αποτελεσματικότητα όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια, πάνω απ' όλα θα πω το εξή. Αυτό θα συμβεί, αυτή η αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα, αυτή η συνοχή θα υπάρξει μόνο αν υπάρχει διαφάνεια και λογοδοσία δεν πρόκειται για κάποια ένωση κάποιων ε, γειτόνων. Είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, δεν μας έχει δείξει το σεβασμό που έπρεπε η Κομισιόν και πρώτη φορά μου πήρε δυόμιση χρόνια να διαπραγματευτώ αυτή την συμφωνία ε, λόγω αυτής της προσέγγισης και της τάσης της Κομισιόν. Και αυτό το λέω κύριε Αντιπρόεδρε, αν η Κομισιόν από δική της βούληση δεν επαστρέψει στο πνεύμα και στις αρχές των συνθήκων, τότε πρόεδρος του Κοινοβουλίου θα πρέπει να τους καλέσει να λογοδοτήσουν και να εξασφαλίσει ότι θα τηρήσουν τις αρχές αυτές. Είναι δικό μας καθήκον να προστατεύσουμε αυτό το θεσμικό όργανο από οποιαδήποτε παρέμβαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Εάν καταφέρετε να κάνετε τελείως ουδέτερη την Κομισιόν, ε, θα, δεν θα έχει τόσο πλάκα πια υπόθεση. λοιπόν, η Κομισιόν έχει τώρα το λόγο. Αγαπητέ Πρόεδρε. Πρόεδρε, αγαπητοί κυρίε και κύριοι βουλευτές, η συζήτηση τώρα έρχεται σε μια στιγμή όπου ολοκληρώνεται μια μακρά και δυσχερή διαδικασία, σημαντικές νομοθετικές τροπολογίες που αφορούν μια πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Υπουργείο 2009 για τη στήριξη των αναπτυσσομένων χωρών μαζί με το μέσον που αφορά τι βιομηχανισμένε και πλουσιότερε χώρε, με το μέσον δηλαδή τη CI. Και έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα για διαδικασίε για συνεργασία στην ανάπτυξη ε, πράγμα το οποίο δεν είχαμε τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε μέσα από την συνήθη αναπτυξιακή βοήθεια. Επίσης προτείνονται μέσα συνοδευτικά της συμφωνίας για το εις ε, διαπραγματεύσεις, για τις εμπορικές διαπραγματεύσεις στο γύρο της Γενέβης, του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου. Και εδώ λοιπόν έχουμε και το μέσο, του μηχανισμό για την μπανάνα, το BAM. Αύριο θα ψηφίσει το Κοινοβούλιο στην δέσμη των τροπολογιών για το μέσον ε, συνεργασίας για την ανάπτυξη για το μέσον που αφορά τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου και για το DCI+. ICI+. Οι διαπραγματεύσει είχαν να κάνουν με πολύ περίπλοκα ζητήματα ω προ τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη θέση ισχύ τη συνθήκη Λισαβόνα. Παρά τι διαφορέ απόψεων που εκδηλώθηκαν μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φρονεί πω έχουν επιτύχει τα θεσμικά όργανα μια ισορροπημένη συμβαστική λύση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δει οι συνάδελφοι κυρία Άστον και κύριο Πίμπαλξ θα ήθελα να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους προς τις δύο πλευράες ε, για τις προσπάθειες που κατέβαλαν στην επιτεύξη μιας συμβαστικής λύσης. Επίσης προς τον Αντιπρόεδρο κύριο Βιντάλ Κουάντρας και τα μέλη της Επιτροπής σας καθώς και προς τις ε, διαδοχικές προεδρίες του Συμβουλίου που οδήγησαν στην συμφωνία υπό την Πολωνική Προεδρία. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εάν αποτύχει αυτή η δέσμη, ε, θα οδηγηθούμε σε πολύ εσφαλμένες λύσεις. Δεν υπάρχει επιλογή δηλαδή αποτυχίας. Θα είναι σημαντικότατο πλήγμα για την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως εμπορικού εταίρου και ως αξιοπιστού αναπτυξιακού εταίρου. Επίσης, δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία σε τομείς κλειδιά με στρατηγικού εταίρους μας. Ως εκ τούτου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ευπρόσδεκτη την απόφαση για ο βραχυπρόθεσμο επίπεδο μέχρι το 2013 δηλαδή και θεωρεί ότι θα πρέπει να ξεκινήσει αμέσως η υλοποίηση του προϋπολογισμού για το ICI Plus και τις πρωτοβουλίες του και τα συνδευτικά μέτρα και την Πανάνα. Ως εκ τούτου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ευγνώμων για την έγκριση του κανονισμού 6-2011-18-19 από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Εάν μπορέσουμε λοιπόν να την υλοποιήσει αυτή το ταχύτερο δυνατό, θα έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα βελτιώσουν την απήχηση των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο και βέβαια θα μπορέσουν να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις σε επίπεδο Γενέβης ε, που, που προκύπτουν από την προσπάθεια για επίλυση μακροχρόνων διαφορών στο θέμα της μπανάνας. Επιτρέπεται δε από τη συμφωνία αυτή περισσότερη διαφάνεια ως προς τις ε, δημοσιονομικές δεσμεύσεις μακροπρόθεσμα. Ταυτόχρονα γίνεται σεβαστή με τη συμφωνία αυτή και η θέση του Συμβουλίου ότι θα πρέπει στην νομοθεσία να συμπεριλαμβάνονται συγκεκριμένες πιστώσεις ή κατανομή πιστώσεων για ορισμένες χώρες ή περιφέρειες. Ιδιαίτερα για τα συνοδευτικά μέτρα της Πανάνας. Το συμβαστικό μέτρα κείμενο ε, ορίζει τρία κριτήρια που θα πρέπει να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον προσδιορισμό των πιστώσεων ανά χώρα. Και έτσι περιλαμβάνει επίσης και μία ένδειξη για τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόζονται τα κριτήρια αυτά. Επίσης συμπεριλαμβάνεται και μια ειδική μνήα για τον τροπο με τον οποιο θα εφαρμοζονται τα κριτηρια αυτα επισης περιλαμβάνεται και μια ειδικη μνηα για προθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταθέσει μια απόφαση υλοποίησης από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ενδεικτικές πιστώσεις χώρα, που θα δίνει στο Συμβούλιο αλλά και το Κοινοβούλιο την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους για τις πιστώσεις αυτές. Τα συνοδευτικά μέσα για τα οποία διατυπώνονται οι υποσχέσεις αυτές μέσα στην ε, Συμφωνία για το Εμπόριο της έχουν μεγάλη σημασία για τις χώρες ΑΚΕ έχουν αρχίσει ήδη οι δασμολογικές περικοπές να αποφέρουν αποτελέσματα και έτσι χρειάζεται αυτή η πρόσθετη βοήθεια για τα κράτη αυτά. Και εν τέλει θα ήθελα να υπενθυμίσω στο Κοινοβούλιο ότι τα κονδύλια που έχουμε υποσχεθεί στα κράτη ΑΚΕ που παράγουν ε, την μπανάνα μέσα από το γύρο της Γενέβης θα πρέπει να είναι συμπληρωματικά και όχι να αντικαταστήσουν το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο. Επίσης, μια και είμαστε στα τέλη του χρηματοπιστωτικού μέσου για την ανάπτυξη, δεν έχουμε άλλο περιθώριο, πρέπει να σας πω, για παράταση αυτού του μέσου. Λίγα λόγια τώρα για το ICI+. Στο ICI+, έχουμε ελάχιστα ποσοστά για τρεις τομείς προτεραιότητας, τη δημόσια διπλωματία, την οικονομική εταιρική σχέση και τις ε, ε, σχέσεις μεταξύ των πολιτών πρόσθετο ποσό για διοικητικές δαπάνες έχει περιληφθεί στο κείμενο. Τα τέσσερα αυτά λοιπόν ποσοστά συνολικά είναι χαμηλότερα από το 100% και άρα επιτρέπουν ένα περιθώριο σημαντικό για ε, διαμόρφωση των ε, συγκεκριμένων ποσοστών των πιστώσεων κατά τη λειτουργία του κανονισμού αναλόγως ε, των αναγκών, της ανάπτυξης στην κάθε περίπτωση και στην κάθε περιοχή και χώρα. Ταυτόχρονα αυτό σημαίνει και συμμετοχή των δύο συνομοθετών στις προτεραιότητες του ICI+. Και για να ολοκληρώσω, Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσβλέπει στην τελική έγκριση της δέσμης από το Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε. Και τώρα στρέφομαι στους ομιλητές εξ ονόματος των ομάδων. Πρώτος είναι ο κύριος Πόγκα. Δύο λεπτά έχετε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αύριο θα αποφασίσουμε για τρίτη φορά για το νέο μέσο συνεργασίας, αναπτυξιακής συνεργασίας που προβλέπει συνοδευτικά μέτρα στον τομέα της μπανάνας για τις χώρες ΑΚΕ παραγωγούς μπανάνας. Μετά από την μείωση της προτιμησιακής ε, ε, δασμολογικής μεταχείρισης στο ΠΑΜΑ. Πρόκειται για 10 χώρες ΑΚΕ μέχρι το 2013. Είναι πολύ μεγάλη σημασία για τους Αφρικανούς εταίρους μας και τους εταίρους της Καραϊβικής στον βαθμό που ο τομέας της μπανάνας έχει μέγα βάρος στις οικονομίες των χωρών αυτών εάν οι δικές μας προτάσεις για τις κατεξοδότητες πράξεις δεν έγιναν δεκτές, ε, είναι πολύ λυπηρό. Ωστόσο, καταφέραμε να κάνουμε κάποια πρόοδο. Το κείμενο προβλέπει σαφείς στόχους, συγκεκριμένα κριτήρια για την κατανομή των πόρων και η Κομισιόν έκανε επίσης μια δήλωση διευκρινίζοντας τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιήσει. Επιπλέον, έχουμε μια δήλωση του Συμβουλίου για το επόμενο δημοσιονομικό, δημοσιονομικό πλαίσιο που διευκρινίζει ότι αυτό θα λάβει καταλήλως υπόψη της κατεξοδότηση πράξης στα μέσα εξωτερικής βοήθειας μετά το 2013. Τέλο, στο ψήφισμά του το Κοινοβούλιο διευκρινίζει και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για προηγούμενο. Και θα πρέπει να σα πω ότι επανέρχομαι το ΤΟΚΟ όπου γινόταν η 22η σύνοδος της ε, Ισομερούς Κοινοβουλευτική Συνέλευση και Ένωσης και θα, και θα σας πω ότι οι Αφρικανοί βασίζονται σε εμά γιατί τα χρήματα αυτά έπρεπε να έχουν απελευθερωθεί πριν από δύο χρόνια. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιε είναι οι εξωθρύνεται συνέπειες για τους εταίρους μας ε, της ΑΚΕ αν απορριφθεί αυτό το σχέδιο ΜΠΑΜ. Η κατάσταση πολλών παραγωγών είναι ε, κρίσιμη και βασίζονται σε αυτό. Ε, και γι' αυτό σας στηρίζομαι σε εσά για να στηρίξετε αυτό το κείμενο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει Πρόεδρος. Και τώρα στρέφομαι στον κύριο Χάουιτ που έχει ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. ότι ασχολούμαστε με την νομιμότητα των ε, κανονισμών, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι συζητάμε το 10% του ευρωπαϊκού προπολογισμού που δαπανάται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στι σχέσει με τον υπόλοιπο κόσμο και για το συμφέρον μα και για την προώθηση των ε, ευρωπαϊκών αξιών για να προστατευτούν οι αδύναμοι του κόσμου πολύ συχνά, σε, χωρίς να το θέλουν αυτό, οι κυβερνήσεις. Θα ήθελα να προσθέσω για τα θέματα νομιμότητας δύο πράγματα. Ότι υποστηρίζω τους συναδέλφου Λόχ και Γκάλ, που είπαν ότι στον πυρήνα των διαθεσμικών συμφωνιών θα πρέπει το, ε, να υπάρχει συναπόφαση στις στρατηγικές αποφάσεις ε, συμπεριλαμβανομένων τέτοιων πιστώσεων με ελάχιστα ποσοστά. Αυτά θα πρέπει να να τηρούνται και κατά δεύτερον ότι και πριν και μετά το 2014 θα πρέπει να ξεκινήσουμε έναν ε, στρατηγικό διάλογο μεταξύ Κοινοβουλίου και σε Επιτροπής για το DHIR για τα άτομα που εμπλέκονται αν ε, δημοσιευθούν ε, και κοινοποιηθούν ε, αυτά τα συμφέροντα, μπορεί αυτό να απειλήσει τη ζωή τους. Ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκφράσει την άποψη ότι θα συνεχιστούν τα όσα ίσχυαν ως σήμερα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα να στραφώ στην κυρία Γκρέζ. Ενάμιση λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, μου το επιτρέπετε αυτή την ε, φράση, οι κατεξιδότητε πράξεις δεν είναι πολύ ελκυστικέ, αλλά είναι πολύ βασικέ. Θα ήθελα καταρχήν να χαιρετήσω την, ε, την εργασία του κ. Γκέρενς ε, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων που δόθηκαν, των αρμοδιοτήτων που δόθηκαν από την συνθήκη της Λισαβόνα σε αυτό το σώμα. Φυσικά και είμαστε υπέρ ε, των συνοδευτικών μέτρων για την μπανάνα, αν και πρέπει να θυμίσουμε ότι η αποζημίωση δεν πρόκειται να λύσει τα προβλήματα των μικρών παραγωγών απέναντι στην Λατινική Αμερική σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά, τη λήψη ισότιμων, ισών δίκαιων μέτρων στον ε, ΠΟΕ. Ωστόσο, αντίθετα, η ομάδα μας είναι αντίθετη, κάθετα αντίθετη, στο να εγκαταλείψουμε τα δικαιώματα που μας δίνει η συνθήκη της Λισαβόνας. Το Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα ε, να βλέπει τι θα γίνει με αυτά τα 180 εκατομμύρια που θα δοθούν και δεν ε, μπορεί να τα αφήσει αυτό στην Κομισιόν στα κρατημέλη. Σας καλώ να απορρίψετε τη συμβιβαστική στη, για το χρηματοδοτικό μέσο DCI BAM που στην ουσία σημαίνει ότι εμείς οι ευρωβουλευτές στην ουσία σαμποτάρουμε εμείς οι ίδιοι τις αρμοδιότητές μας. Σας ευχαριστώ. Και τώρα στρέφομαι στον κύριο Μέγερ. Για ένα λεπτό έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Βιδάλ Κουάδρας, αναγνωρίζω ότι πράγματι μπορέσατε να αλλάξετε άρδιν την αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να μην βρίσκεται στην, ε, σε αμφιβολία ως προς τη συναπόφαση στις διαδικασίες αυτές. Ξέρω ότι είναι πολύ επικριτική η ομάδα μου ως προς το ε, DCI δεν μπορούμε να ορίζουμε το, για το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου δεν μπορούμε δηλαδή να ορίζουμε ότι κάποια δικαιώματα είναι πιο σημαντικά από άλλα ή ότι ισχύουν κάπου αλλά δεν ισχύουν κάπου αλλού τα είδαμε αυτά και με την περίπτωση του Καντάφη και με τόσες άλλες Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε περισσότερο τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και κατά τα άλλα ξέρω ότι έχετε δουλέψει πολύ και κάνατε και όλους τους άλλους να δουλέψουν μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ακούμε εκ μέρους... Έχουμε τώρα τον κύριο Λίζεκ για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρίε και κύριοι συνάδελφοι. Επιτρέψτε μου δύο λόγια για να επικεντρωθώ στο νομοθέτημα που αφορά το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου δηλαδή δημοκρατία, πολιτική εκπροσώπηση, δημοκρατική εκπροσώπηση, ανθρώπινα δικαιώματα και που επιτρέπει να παρεμβαίνουμε σε πάρα πολύ δύσκολε πολλέ φορέ περιστάσει. Γιατί μπορεί να ζούμε στον 21ο αιώνα, αλλά βλέπουμε ακόμη πολύ συχνά βασανιστήρια, διώξει, εκμετάλλευση σεξουαλική των παιδιών και πολλά άλλα δεινά. Βέβαια, δεν μπορούμε να σώσουμε όλο τον κόσμο μέσα από το μέσο αυτόν, αυτό, αλλά μπορούμε ή μη τι άλλο να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη τη κοινωνία των πολιτών, στην προαγωγή του ε, δικαιώματο στην ελεύθερη έκφραση, στο δικαίωμα τη ελευθερωτυπία, στα ελεύθερα μέσα μαζική ενημέρωση. Και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο εκ τούτου. Ε, επιτρέψτε μου να παραθέτω και την ε, γνωστή ταινία Nobody's Perfect. Κανεί δεν είναι τέλειο. Ε, λοιπόν, αυτό που μα έχει μείνει πλέον ω εναλλακτική είναι να δεχθούμε ή να απορρίψουμε αυτό το μέσο. σω κάποια στιγμή μπορέσουμε να ενισχύσουμε τη θέση του Κοινοβουλίου, αλλά τώρα πρέπει να εγκριθεί. Ο πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ κύριε Λίσσα και κυρία Γκόμε για ένα μισή λεπτό. Uh, Πρόεδρε, με χαρά αναγνωρίζω ότι όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, έχουμε ήδη μια διαδικασία ανάμεσα σε εμά και την Κομισιόν που μας επιτρέπει τον έλεγχο Χρειάζεται να αναπτυχθούν διαδικασίες που να είναι ευέλικτες και γνωστές, ιδιαίτερα για τις, μέσω των αντιπροσωπιών μας επιτόπου που πρέπει να εργαστούν περισσότερο ενημερώνοντας οργανώσεις, ΜΚΟ και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κτλ. Επίσης θα πρέπει να βλέπουμε τι συμβαίνει με την εφαρμογή των προγραμμάτων, ενώ υποτίθεται πως το μέσο αυτό προστατεύει του οργανισμού αυτού τις ενώσει και του ανθρώπου. Επίση, θα πρέπει να βοηθήσουμε να αποφευθεί η λογοκρισία και κυρίω η λογοκρισία στο ίντερνετ. Αλλά α μιλήσω για την κατεξουσιοδότηση, πράξη κατεξουσιοδότηση πράξης και για το DCI. Εγώ λυπούμαι για την τακτική, την εκβιαστική που χρησιμοποίησαν το Συμβούλιο και η Κομισιόν ώστε να προσπαθήσουν να κάνουν αυτό το Κοινοβούλιο να ε, παραδώσει τις αρμοδιότητες που του έχουν δοθεί μέσω της συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν μπορεί το Κοινοβούλιο να εγκαταλείψει αυτές τις αρμοδιότητες. Είναι υποχρέωσή του να ασκεί τον δημοκρατικό έλεγχο σε ένα μέσο όπως το DCI που έχει τεράστιες δυνατότητες για την ανάπτυξη για ολόκληρο τον κόσμο. Δεν δεχόμαστε αυτό το είδο τις τακτικές ούτε τις απειλές ε, ε, που έγιναν γιατί δεν θα τηρήσουμε υποτίθεται τις υποχρεώσεις μας ε, για το χρηματοδοτικό μέσο για την μπανάνα. Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε. Ευχαριστούμε κυρία Γκό μα. Η κυρία Κολάσκα Μπομπίνσκα για δύο λεπτά τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επιτροπέ. Λυπάμαι που το Κοινοβούλιο δεν μπόρεσε να προσπιστεί πλήρω τη θέση του κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υποστηρίζω την ε, θέση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο μέλλον θα πρέπει να διαδραματίζει μεγαλύτερο ρόλο για το πώς δαπανώνται οι πόροι υπό το μέσο αυτό οι αιρετοί θα πρέπει να αποφασίσουν τα πράγματα αυτά και όχι οι ομάδε εργασία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα σημαντικά αυτά θέματα. Παρά το γεγονό αυτό, θα υπερψηφίσω το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Μέσο για την Πραγωγή τη Δημοκρατία και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, γιατί θεωρώ ότι το μέσο αυτό είναι είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν θα πρέπει να τύχη περαιτέρω καθυστέρηση. Θα πρέπει να προάγουμε τη δημοκρατία στη Ρωσία, στο Ιράν, στην Ουκρανία. Πρόεδρε, θα πρέπει σήμερα να διευρύνουμε τις ε, δράσεις μας στους τομείς αυτής. Πέρα από το χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας, θα πρέπει να δημιουργηθεί και ένα ευρωπαϊκό ίδρυμα για τη δημοκρατία. Η αρχική ιδέα του Ευρωπαϊκού Χρηματοποιητικού Μέσου για την Πραγωγή της Δημοκρατίας ήταν ακριβώς ένα τέτοιο ίδρυμα. Και τώρα λοιπόν θα πρέπει να λάβει σάρκα και αυτή η ιδέα. Νομίζω ότι τα συνδυασμένα αυτά δύο μέσα θα προωθήσουν την θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη δημοκρατία σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ, κυρία Κολάσκα Μπομπίνσκα. Τώρα ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ο συντονιστής μας, ε, Τζίτερμαν, δεν μπορεί να είναι παρόν ε, για προσωπικούς λόγους. Ωστόσο, συμμερίζομαι απόλυτα την ανάλυση του για αυτό το θέμα. Η διαβούλευση για αυτό το θέμα ήταν μακρά και ε, δύσκολη και αν ε, το μέσο για την ε, δημοκρατία και τα δικαιώματα των ανθρώπων ε, είναι ικανοποιητικό, πολύ λιγότερο συμβαίνει αυτό με τη συμβιβαστική για την μπανάνα. Η εντολή που δόθηκε στην ομάδα τη διαπραγματευτική μας ήταν να τοποθετήσει το Κοινοβούλιο στο ίδιο επίπεδο με το Συμβούλιο για όλες τις αποφάσεις προγραμματικές όσον αφορά την επιλογή των στατικικών επιλογών και τις πρικοδοτήσεις. Γιατί είναι οι αρμοδιότητες αυτού ίδιο του σώματος και το ίδιο το πνεύμα της συνθήκης Λιθαβόνας που διακυβεύονται εδώ. Η επιλογή αυτού του προγραμματισμού είναι μια πολιτική επιλογή όπου το δικό μας σώμα πρέπει να έχει λόγο. Αρνούμενο κατηγορηματικά την αναγνώριση αυτής της αρμοδιότητας, το Συμβούλιο ακόμα μια φορά δείχνει έλλειμμα ιδεολογικό που καταδικαστέο. Ε, θα πρέπει λοιπόν από εδώ και μπρος να δεχτεί πως η εξωτερική αναπτυξιακή βοήθεια είναι κοινή αρμοδιότητα των δύο θεσμικών οργάνων και γι' αυτό και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να δείξει ότι, μέσω αυτό της μπανάνας ότι χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια στις κοινοτικές αποφάσεις. Αν χάσουμε αυτή τη μάχη θα, ε, θα ίσχυε το παράλογο ότι θα πρέπει να περιμένουμε μια νέα συνθήκη για να επιτύχουμε επιτέλους τις ε, εξουσίες τις οποίες ήδη προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας. Ευχαριστώ κύριε Τυρολιά. Και τώρα περνάμε στη δικασία Κατσουδιάη με τον κύριο Προτασίεβιτς πρώτο. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Ως πρόεδρος της αντιπροσωπίας κοινοβουλευτική για τη σχέση με τη Λευκορωσία. Είμαι σε θέση να γνωρίζω πόσο μεγάλη σημασία έχει το μέσο αυτό, το ευρωπαϊκό για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου, ιδιαίτερα για τις χώρες εκείνες όπου ε, επικρατούν ολοκληρωτικά καθεστώτα. Και έχω ένα πολύ ε, λυπηρό παράδειγμα να σας παρουσιάσω. Έναν ε, άνθρωπο ο οποίο καταδικάστηκε σε καταναγκαστικά έργα για πολλά χρόνια στην Λευκορωσία μόνο και μόνο επειδή ήταν αγωνιστής για τη δημοκρατία. Αυτό δείχνει πόσο σημαντικά είναι αυτά τα μέσα. Πρέπει αυτού του ανθρώπους να τους προστατέψουμε από τα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Χαίρομαι που μπόρεσαμε να καταλήξουμε σε αυτέ τι συμβαστικέ λύσει. Είναι πολύ πιο ευέλικτα από ό,τι στο παρελθόν τα μέσα αυτά τώρα. Και ελπίζω ότι στο μέλλον θα έχουμε τη δυνατότητα να στηρίζουμε περισσότερο ακόμη τι οργανώσει εκείνε οι οποίε αγωνίζονται για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε χώρε όπω η Λευκορωσία. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Προτασίευη, τη λέει ο πρόεδρο, ο κύριο Πάσκο. Ευχαριστώ. Στις 9 Απριλίου 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την ε, ε, αλλαγή του μηχανισμού 1934 του 2006 και τότε οι θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ήταν διαφορετικές γιατί ήταν σημαντικό να βρεθεί μια διαδικασία συνδιαλλαγής ε, προκειμένου να προσεγγίσουν οι θέσεις. Εν τω μεταξύ, έγιναν οκτώ τριμερείς ε, διάλογοι και τελικά καταλήγαμε, καταλήξαμε σήμερα να λαμβάνονται αποφάσεις μέσω ε, συναπόφαση και μέσω των ε, πράξεων κατά εξουσιοδότηση ενισχύει το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έτσι αυτό δίνει ελπίδε για την επιτυχή ολοκλήρωση του θέματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Καπάσκα. Η κυρία Μπασέσκου έχει το λόγο τώρα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. σε ό,τι αφορά την τρέχουσα οικονομική κρίση. Είναι σημαντικό το ότι συζητάμε την έκθεση αυτή. Και το σημείο 5 της έκθεσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι εμπορικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να λάβουν και μια γεωγραφική καταδάξη. Είναι σημαντικό οι ευρωπαϊκές Εταιρικέ σχέσεις να ανταποξέλθουν στις σημερινές προκλήσεις, όπως για παράδειγμα η αιρεσιμότητα της υποστηρίξης ε, σε ό,τι αφορά περιβαλλοντικούς όρους ή σε ό,τι αφορά ε, χώρες οι οποίες έχουν μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης αλλά παρουσιάζουν σημαντική καθυστέρηση. Μιλάμε επίσης για την εφαρμογή της συνθήκης του Κιώτο. Οι όροι που ορίζει η Παγκόσμια Οργάνωση Εργασία θα πρέπει να τηρηθούν και τα πολύ θεμελιώδη δικαιώματα δεν μπορούν πολύ απλά να καταπατώνται. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Μπασέσκου. Ο συνάδελφο Σικέσκη. Πρόεδρε, τα μέσα αυτά μας επιτρέπουν ε, να υλοποιήσουμε πολύ σαφείς στόχους ως προς την εξωτερική μας δράση. Στόχους που αφορούν και την αναπτυξιακή πολιτική. Τα μέσα πρέπει να είναι πολύ ρονταρισμένα, πολύ λεπτά σχεδιασμένα ε, και με συγκεκριμένους στόχους για τη δημοκρατία, για την εκπαίδευση, ενδεχομένω το επιχειρήν, την ανθρωπιστική βοήθεια, την ανάπτυξη τη Δημοκρατία, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, όλα αυτά είναι ερωτηματικά που τίθενται. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι όργανο που εκλέγουν οι ίδιοι οι πολίτε και ω εκ τούτου έχει ιδιαίτερα και κατεξοχήν το δικαίωμα να τοποθετείται, να τοποθετείται ως προς την χορήγηση, ω προ την κατανομή των πιστώσεων ε, για την ε, δημοκρατία, για τι ελευθερίε. Η κοινωνία και για την κοινωνία των πολιτών φυσικά, αλλά και για την ολοκλήρωση ε, στόχων που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σικέσκη. Ολοκληρώνεται έτσι η διαδικασία Καρστιάη και παρακαλώ τον κύριο Πίτερ να είναι λόγο. Thank you very much, uh, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η συζήτηση ήταν ε, ενδιαφέρουσα και άνοιξε το δρόμο για περισσότερη κατανόηση και ελπίζω πιο πολύ συνεργασία στο μέλλον. Ως προς αυτό, άκουσα τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου και είμαι βέβαιος ότι θα ανταποκριθούμε σε αυτές στο επόμενο πολυετές ε, ε, δημοσιονομικό πλαίσιο όταν θα το υποβάλουμε στα επόμενες, στις επόμενες εβδομάδες. Συμφωνώ όμως με πολλούς από εσάς που είπαν ότι ακόμα και τώρα χρειάζεται να δοθεί προστασία σε όσους υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Κομισιόν συμφωνεί πως είναι ένα πρόβλημα όπου τα καθεστώτα χρησιμοποιούν ε, τους νόμους για να καταπιέζουν περισσότερο τα φορολογικά, τη φορολογική νομοθεσία για να καταπιέζουν περισσότερο τις ΜΚΟ και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ξέρετε, κύριοι βουλευτές, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι η Κομισιόν είναι ευαίσθητη στα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ήδη ανέλαβε την ε, δέσμευση να ανταποκριθεί πλήρως ε, στις ε, υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συνθήκη της Λισεβόνας. Στην περιστατική για το 2020 κάναμε πράξη αυτή την δέσμευσή μας όσον αφορά τις τη πράξεις και Αναφερθήκατε σε αυτό το τμήμα του κειμένου, δεν χρειάζεται να το παραθέσω εκ νέου, κυρία Μπίλερ. Να σας πω και πάλι ότι η σημερινή συμβιβαστική πρόταση αποτελεί μια ισορροπημένη πρόταση ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Κάθε πλευρά βλέπει πράγματα που ε, τη βρίσκουν σύμφωνοι και άλλα που όχι. Όμως θα πρέπει να ξεπεράσουμε το περιορισμένο πεδίο των ε, διοργανικών σχέσεων. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, όπως δήλωσα στη συζήτηση, το να εγκριθεί αυτό το πακέτο δεν είναι επιλογή. Ε, δεν υπάρχει μάλλον επιλογή, δεν υπάρχει δε plan B. Εάν δεν δεχτεί το Κοινοβούλιο αυτό το σχέδιο, δεν θα έχουμε βάση για να, να εφαρμόσουμε το ICI Plus και τα συνδευτικά μέτρα για την μπανάνα. Με το ICI Plus δεν θα μπορέσουμε να προωθήσουμε τα συμφέροντά μας και το κύριο μας στο εξωτερικό. Για τα συνδευτικά μέτρα για την μπανάνα, η Κομισιόν θέλει να δηλώσει ξεκάθαρα πως δεν υπάρχουν κονδύλια από οποιαδήποτε άλλη πηγή, όπως το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο. Εάν δεν υιοθετηθεί ε, το μέσο για τα συνδευτικά μέτρα για την μπανάνα, ο Ευρωπαϊκή Ένωση θα θεωρηθεί αναξιόπιστος εμπορικός εταίρος και αναξιόπιστη απέναντι στους στοχότερους ε, τέρους μας της Αυτό δεν, το δεν είναι αυτό που αναμένουν οι πολίτες μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, θα ήθελα να επιμείνω για το γεγονός ότι αυτή η συμβιβαστική είναι καλό αποτέλεσμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως έναν ε, ενιαίο παίκτη στην εξωτερική της διάστασης διάσταση τόσο όσον αφορά την ευρωπαϊκή συνεργασία με τους στρατηγικούς της εταίρους αλλά και όσο αφορά τις ε, χώρες ΑΚΕ παραγωγούς μπανάνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ξανακούμε τώρα τους συγητές με τον κύριο Γκέρνς πρώτα, τρία λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μόλις άκουσα τον Επίτροπο κύριο Φίλε, ο οποίος επικαλείται μια καλή συνεργατική δράση μέσα στο Κοινοβούλιο, μέσα στην Ολομέλεια, παραθέτω τα λόγια του. Ευχαριστώ να συνεργαστούμε με ποιον είναι εδώ. Αλλά ποιον είναι εδώ. Γιατί από την άλλη πλευρά του το Συμβούλιο δεν είναι κανένας. Δεν άκουσα ούτε απάντηση, ούτε καμία θέση από πλευρά του Συμβουλίου. Και αν ήταν εδώ παρόν το Συμβούλιο με εκπροσώπου του σήμερα, θα μπορούσαμε ενδεχομένω να αντιπαρατεθούμε τα σημεία στα οποία διαφωνούμε και ακόμα και αυτά στα οποία συμφωνούμε. Ε, πράγμα το οποίο έχω την ευκαιρία να πράξω και στο πλαίσιο τη Επιτροπή Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Φερρυπίν, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ένα κοινό όραμα για τη συνεργασία στην ανάπτυξη για την Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη, στην οποία άλλωστε μα καλεί να αναλάβουμε δράση η συνθήκη τη Λισαβόνα, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να μεταφραστεί και σε κοινέ ευθύνε. Υπογραμμίζω κοινέ ευθύνε. Τι, σημαίνει αυτό τι συμβαίνει όμω τώρα. Συμβαίνει ότι τα κράτη-μέλη δαπανούν υπό δική τους μόνο ευθύνη 80% των ποσών στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας για την ανάπτυξη και είναι Προφανέ ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουν και τελευταία λέξη τα κράτη-μέλη όσον αφορά του εθνικού του προπολογισμού και, και το Κοινοβούλιο δεν έχει λόγο, ούτε αντίρρηση. Από την άλλη όμως εμπιστεύονται ένα σημαντικό ποσό στην, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα κράτη-μέλη, το οποίο αυτή διαχειρίζεται με βάση την εντολή που τη χορηγούν τα κράτη-μέλη, δηλαδή το Ταμείο για την Ανάπτυξη. Και όσο δεν υπάρχει αυτή η ε, κοινή διαχείριση, το κοινοβούλιο θα μένει πάντα στο περιθώριο. Δηλαδή θα έχει καλυφθεί το 9% των ποσών που πάνε στην ανάπτυξη. Και μετά υπάρχει ένα ελάχιστο ποσό που αποδίδεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για Διαχείριση και στο οποίο μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επικαλέσει το άρθρο 291 και όπου είναι ισότιμο συνομοθέτη με το Συμβούλιο, όπου και πάλι το Συμβούλιο θέλει να μα βάλει στο περιθώριο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Θέλουμε το Κοινοβούλιο να παίξει τον ρόλο που του αναλογεί στο πλαίσιο τη ανάπτυξη μια πραγματική ε, πολιτική συνεργασία για την ανάπτυξη. Φαίνεται ότι δεν έχει καταλάβει ε, το μήνυμα το Συμβούλιο και απαιτεί και στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση και το τελευταίο αυτό ε, αναλογικό ποσό το Συμβούλιο να μείνει το Κοινοβούλιο στο περιθώριο. Άλλωστε αυτό έχει προσπαθήσει να πράξει και υπό Ουγγρική Προεδρία το Συμβούλιο και το θυμόμαστε πάρα πολύ καλά γιατί αφενός λέει ε, απευθύνει έκκληση για, για συνεργασία, πολιτική συνεργασία, αφετέρου όμως δεν μας χορηγούνται καν μέσα τα οποία θα μας επέτρεπαν να συνεργαστούμε και θα μας επέτρεπαν να συμπεριφερθούμε με κάποια εν περιπτώσει αξιοπρέπεια έναντι των θεσμικών μα εταίρων. Το Κοινοβούλιο όμω δεν εσώπασε όταν ήταν η εποχή όπου βρίσκονταν σε δύσκολη θέση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έπρεπε να ενσωματωθεί το χρηματοπιστωτικό μέσο για την ε, ανάπτυξη ε, στην, ε, στο μέσο για την εξωτερική δράση δεν εφίστημε ουδενίας προσπάθειας και κόπου για να σας βοηθήσουμε κυρία Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεπάρξετε με τη νέα ύπατη εκπρόσωπος προς την για την εξωτερική πολιτική όταν ήταν δύσκολες εποχές για σας και νομίζω ότι η μη τι άλλο οι προσπάθειες οι οποίες ε, κατέβαλε το Κοινοβούλιο και δι' η Επιτροπή Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η μη τι άλλο θα άξιζαν θα άξιζαν αντίστοιχη συμπεριφορά και πιο ορατή συμπεριφορά από τα θεσμικά όργανα. Από τα άλλα θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Γκέρενς. Ο κύριος Σόλτς. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε κύριε Επίτροπε. Η κριτική προς το Συμβούλιο με βρίσκει σύμφωνο και συμφωνώ με τον συναδελφό Γκέρενς. Ε, θα ήθελα να πω κλείνοντας τη συζήτηση ότι μετά από όλες τις κουβέντες που ακούσαμε για τις διαπραγματεύσεις, του συμβιβασμού κτλ να πω ότι θεωρώ ότι υπάρχει ε, ένα καθήκον, μια εργασία σε ό,τι αφορά το δικό μου μέσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτήσει ένα έγγραφο ε, στρατηγικής για το ICI+. Δεν μπορούμε ως νομοθέτες ε, να αφήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει με ένα παλιό έγγραφο το οποίο καταρτίστηκε πριν από την αλλαγή των αρμοδιοτήτων. Οι νομοθετές έχουν δώσει μια νέα όθηση σε ό,τι αφορά την προσέγγιση ε, προς τους εταίρους και άλλοι κεντρικοί πολιτικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στήφονται στο επίκεντρο σε ό,τι αφορά η συνοχή, η τήρηση των διεθνών προτύπων, σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση των περιβαλλοντικών στόχων, αλλά το έγγραφο στρατηγικής ε, αγνοεί αυτούς τους στέχους και μέσω το μέσο αυτό αναφέρεται ότι θα πρέπει να άρει εμπόδια σε ό,τι αφορά την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είχαμε αυτό υπόψη ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλαμε όχι ένα εργαλείο κατάληψης, αλλά ένα εργαλείο συνεργασίας. Θέλουμε λοιπόν στο μέλλον να έχουμε στρατηγική έγγραφα στρατηγικής. Δεν θέλουμε να γράφουμε εμείς. Αυτό το έχουμε πει πολλέ ε, φορές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να το κάνει αυτό, αλλά θέλουμε δικαίωμα βέτο σε περίπτωση που αγνοούνται οι προδιαγραφέ που έχουμε ορίσει. Γι' αυτό λοιπόν ε, οι προτάσει για τις νέες γενιές ε, χρηματοδοτικού μέσου θα πρέπει να χρησιμοποιούν με καλό τρόπο τις καταξιοβιώτες πράξεις. Ευχαριστώ πολύ και τώρα η κυρία Γκάλ για δύο λεπτά έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να θα ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο. Θα ήθελα να τονίσω ότι κατανοώ απόλυτα τους συναδέλφους εκείνους οι οποίοι θεωρούν ότι στο σημείο αυτό μπορεί να, τεθεί να και να δημιουργηθεί ένα προηγούμενο Θέλουμε να υπάρχουν αποτελεσματικά και αποδοτικά, χρηματοδοτικά μέσα τα οποία θα εκπληρώνουν το σκοπό τους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την πραγωγή της δημοκρατίας και των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χρειαζόμαστε μία κοινή στρατηγική, η οποία θα πρέπει να διατυπωθεί με τον πολίτη, με συνεργασία με τον πολίτη. Οι πολυετής ε, στρατηγικές προφανώς δεν μπορούν να αποφασιστούν χωρίς την συμμετοχή του πολίτη. Είναι ακατανόητο και πικρό αν θέλετε. Δυσκολεύομαι να καταλάβω γιατί ε, προβάλλουν αντίσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταλαβαίνω λοιπόν την στάση των συναδέλφων. Θα πρέπει να δούμε ωστόσο ότι καταλήξαμε σε ένα συμβιβασμό ότι κάναμε παρόλα αυτά ένα βήμα προς τα εμπρός σε ό,τι αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα. Και έτσι θα πρέπει να αντιληφθούμε το βήμα αυτό, σε ένα βήμα προς τα μπροστά. Αναμένουμε όλα όσα αποφασίστηκαν να πραγματοποιηθούν στην επόμενη δημοσιονομική περίοδο. Και είναι διτό το έργο μας. Είναι διτή η ευθύνη που φέρουμε. Γιατί ο αγώνας αυτός ε, έχει πάρει ήδη δύο χρόνια και εμείς θα πρέπει να, να σταθούμε στο ύψο των περιστάσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο πρόεδρο Και τώρα δύο λεπτά η κυρία Λόχπιλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και επιτρέψτε μου να επανέλθω στο μέσον για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα των ανθρώπων. Δείχνει η συζήτηση ότι το μέσον αυτό είναι μέσο στο οποίο πάντοτε στηρίζει πολλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ταυτόχρονα όμω και με το Ευρωπαϊκό Κληροδότημα Καταπίστευμα για τη Δημοκρατία, ε, βλέπουμε την ανάγκη να είναι πολύ πιο ευέλικτο αυτό το μέσο, να μπορεί να ε, στηρίξει ταχαίως ε, κατεπηγόντω υποθέσει που έχουν να κάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα με κυβερνητικέ οργανώσει κ.ο.κ. Επιτρέψτε μου όμω και να αναφέρω το εξή για άλλη μια φορά, ότι η αρχή ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρεμβαίνει στη διαμόρφωση, τη λειτουργία, την ε, κατανομή των πόρων αυτού του μέσου έχει γίνει αποδεκτό από όλε τι πλευρέ, τόσο τα θεσμικά όργανα όσο και την κοινωνία των πολιτών. Και γι' αυτό παρακαλώ του συναδέλφου να ανασκουμποθούν για την προσεχή μάχη που μα περιμένει. Γιατί είχαμε πολεμήσει για τη σύσταση του, του ίδιου του μέσου. Τώρα πρέπει να αγωνιστούμε για τη βελτίωσή του. Σα ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ και την κυρία Λόχπιλος. Και τώρα ο κύριος Μίτσελ δύο λεπτά. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και καταρχάς ευχαριστώ τον κύριο Βιδάλ Κουάντρας για τις προσπάθειές του στη διαδικασία της συνδιαλλαγής και ότι παραμένουν αρκετές α, επιφυλάξεις. Ξέρω πολύ καλά ότι ο ίδιος έκανε ό,τι μπορούσε για να επιφέρει την ε, καλύτερη δυνατή συμβαστική λύση υπό τις δεδομένες συνθήκες. Πλην όμω και του η συνθήκη της Λισαβόνας, για την οποία η πατρίδα μου διεξήγα και δύο δημοψηφίσματα, προβλέπει συναπόφαση μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σε διάφορους τομείς, μεταξύ των οποίων και η συνεργασία για την ανάπτυξη. Και δεν βλέπω να συμβαίνει αυτό τώρα. Όπου δηλαδή συμμετέχει στην ενλήψη αποφάσεων σε νομοθετική διαδικασία το Συμβούλιο, θα πρέπει να συμμετέχει εξίσου και το Κοινοβούλιο. Εγώ αυτό δεν το βλέπω. Ούτε στη μικροδιαχείριση να συμβαίνει, ούτε βλέπω να υπάρχει η δυνατότητα, τα μέσα, ο χρόνο για να εξασφαλιστεί αυτό. Αλλά είναι ευθύνη μα, καθήκον μα και μάλιστα εξουσία απορρέουσα από τη συνθήκη να το διεκδικήσουμε. Όταν ήμουν μικρός λέγανε ότι είσαι αυτός, αυτό που κάνεις. Δεν μπορούμε να λέμε το ένα πράγμα και μετά να κάνουμε το άλλο. Και λέμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκάθαρα ότι αυτό που πράττει σε σχέση με τις εξουσίες, με και τον διαχωρισμό εξουσιών μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την ανισομερή, ανισομερή κατανομή είναι πολύ απογοητευτικό. Και ξέρω ότι θα έρθει η ώρα που θα έρθει να χτυπήσετε την πόρτα του Κοινοβουλίου και σα διαβεβαιώ ότι το Κοινοβούλιο δεν θα σα ανοίξει τι αγκάλε του όπω θα περιμένατε ενδεχομένω. Για δε το μέσον στο οποίο εγώ έχω ιδιαίτερα η ε, ευθύνη στη σύνταξη εκθέσεων του μηχανισμό, δηλαδή χρηματοδότηση αναπτυξιακή συνεργασία, δεν θέλω να πω ότι αυτά τα 6 δι έτος ε, που αναφέρθηκαν και από τον κύριο Επίτροπο, βεβαίω και θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν ε, την διάσωση πάρα πολλών ανθρώπινων ζωών, εφόσον έχουμε επαρκή συνοχή. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μίτσλ και τώρα παρακαλώ τον κύριο Βιντάλ Κουάντρας να λάβει το μέρος ως συντονιστή της αντιπροσωπείας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να κλείσω με μια υποκειμενική παρατηρήση. Ως Πρόεδρος ε, και επικεφαλής μάλλον των διαπραγματεύσεων αυτών, αισθάνομαι ως σαν καθηγητής και σαν φοιτητής. Ε. όπου τελικά ο φοιτητής ε, κατσαδιάζεται παρόλο που τα έκανε όλα τέλεια σχεδόν. Όλα τα βασικά στοιχεία του μέσου αυτού περιλαμβάνονται ε, σε αυτή την ενδιάμεση συμφωνία στην συναπόφαση. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό μήνυμα για το μέλλον. υπήρξε πολιτική δήλωση για δέσμευση, για πλήρη χρήση των ε, κατεξουσιοδότηση πράξεων ε, στο μέλλον, σε τέτοιου είδου μέσα. Άρα, όταν συζητάμε στρατηγικά ζητήματα, θεωρώ ότι από στρατηγική άποψη ε, με τη συμφωνία αυτή κάναμε ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Ασφαλώς, όταν κάθεται κανείς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συζητήσει κάθε μία χώρα που εξάγει μπανάνες και το πώς θα ταπανηθούν τα κονδύλια που χορηγούνται στη χώρα αυτή ευρώ προς ευρώ και σύμφωνα με τις διάφορες ε, προτεραιότητες και τα διάφορα κριτήρια, ε, στη φάση αυτή ασφαλώς θα έχουν να πούν κάτι τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο των προηγούμενων διαδικασιών, αλλά θεωρώ αν ζητήσουμε από τα κράτη -μέλη, αν ζητήσουν τα κράτη-μέλη να εξαιρεθούμε από την διαδικασία αυτή, νομίζω ότι πραγματικά τι να πω. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε λοιπόν ότι σημειώσαμε πρώτο. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι πολιτικέ και κοινωνικέ συνέπειε μια αποτυχία στην παρούσα φάση θα ήταν πραγματικά ανυπολόγιστε. Άρα, επαναλαμβάνω την θέση μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, ε, ολοκληρώνεται λοιπόν η κοινή συζήτηση. Αύριο στις 12 θα διεξαχθεί η ψηφοφορία. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη ε, είναι η δήλωση της Επιτροπής για το Φόρουμ Ενιαίας Αγοράς.